δεν χρειάζεται το Κοινοβούλιο να δραστηριοποιηθεί στην παρούσα φάση της διαδικασίας. Λαμβάνει ε, γνώση το Κοινοβούλιο και θα ενημερώσει τις αρμόδιες ρουμανικές αρχές. Από ε, τις ομάδες EFTD, EFN και ECR έχω λάβει αιτήματα για διορισμούς και αλλαγές σε επιτροπές και κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες. Στα πρακτικά θα βρείτε τους καταλόγους αυτούς και αν δεν διαφωνείτε